ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Η συζήτηση τελείωσε. Η ψηφοφορία αύριο στις 12 η ώρα. Επόμενο θέμα. Έκθεση της κυρίας Κλέβα και εφαρμογή και αντίκτυπο των μέτρων για την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή. Και θα ήθελα να ακούσουμε τώρα την κυρία Σιγητρέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους και οδησίγητες για την εξαιρετική συνεργασία στους τελευταίους μήνες. Η αποτελεσματική χρήση της ενέργειας είναι βασικό μέρος της στρατηγικής 2020. Η Ευρώπη έχει πάρα πολλά να κάνει πώς να μειώσει την συνολική κατανάλωση ενέργειας κατά 20% μέχρι το 2020. Γι' αυτό θεωρώ πως όλες οι σχετικές πολιτικές όπως η πολιτική συνοχής πρέπει να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο. Με την έκθεσή μου θα ήθελα και πάλι να τονίσω τα ωφέλη της ενεργειακής αποδοτικότητας η οποία μπορεί να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά μας ε, να οδηγήσει σε πράσινη ανάπτυξη και περισσότερες δουλειές. Οι επενδύσεις επίσης είναι μια ευκαιρία να καταπολεμήσουμε την οικονομική κρίση και την κλιματική αλλαγή. Η ανάλυση των υφιστάμενων μέτρων δείχνουν πως οι βασικοί αρνητικοί παράγοντες είναι η ανεπαρκής ενημέρωση, η ανεπαρκή οικονομικά κίνητρα, το χαμηλό προφίλ του θέματος αυτού και ανεπαρκής εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας. Είναι λοιπόν σαφές πως στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2007-2013 ε, τα προβλήματα είναι περισσότερο πρακτικά και όχι νομοθετικά. Στο πλαίσιο λοιπόν των συμφωνημένων αλλαγών στο νομοθετικό πλαίσιο της ε, πολιτικής συνοχής έχουμε συγκεντρώσει πολλές διαφορετικές προτάσεις στην έκθεση για το πώς ε, θα συμπεριληφθεί η ενεργειακή απόδοση στον επόμενο προϋπολογισμό. Είναι λοιπόν από τα βασικά εργαλεία που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη διάθεσή της για να βελτιώσει την ευρωπαϊκή οικονομία και να διασφαλίσει υψηλότερη ενεργειακή αποδοτικότητα. Είναι σημαντικό τα κράτη-μέλη να θεωρήσουν τη χρηματοδότηση αυτή ως ε, επένδυση και ως ευκαιρία. Η κατανομή κονδυλίων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης θα διασφαλίσει μακροπρόθεσμο προγραμματισμό για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στο πλαίσιο της οικονομικής ε, ανάκαμψης και των ε, περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων των ΟΤΑ πρέπει να φροντίσουμε οι οργανισμοί τουρκικής αυτοδιοίκησης ε, να έχουν περισσότερες δυνατότητες χρηματοδότησης. Πρέπει να φροντίσουμε πως όλα τα επίπεδα της διοίκησης ε, θα εμπλακούν στο εθνικό, τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, στο πλαίσιο της ε, ενεργειακής απόδοσης, να υπάρξει συντονισμός με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα μέτρα λιτότητας βεβαίως καθιστούν δύσκολο για τα κράτη-μέλη να συγχρηματοδοτήσουν ε, τα προγράμματα αυτά. Γι' αυτό είναι σημαντικό να βρούμε νέους καινοτρόμους τρόπους χρηματοδότησης. Είμαι σίγουρη πως πρέπει εδώ πέρα να συνδυαστούν επιδοτήσεις με άλλα χρηματοδοτικά μέσα για να δημιουργηθούν νέες ΣΔΙΤ και να έχουμε νέες επενδύσεις. Η Κομισιόν ήδη έχει εργαστεί προς αυτή την κατεύθυνση. Προς την κατεύθυνση δηλαδή συγκεκριμένων προτάσεων και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να απολυμήσουμε την ενεργειακή φτώχεια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Δύο συναδελφοί έχουν ζητήσει τον λόγο. Ο κύριος Μπάνκη. Θέλω να σας δώσω τη στρατάλη που τη στρατική επισηρωτάσω. Ενώ είναι φόντος γέραντης ο Σούχησεν, ο Ζένεργη Χατήκοησέγ, ο Ζέρουπαϊκού. Ευχαριστώ πολύ. Πρόκειται για μια πάρα πολύ σοβαρή έκθεση, ουσιαστική έκθεση. Είναι σίγουρο ότι δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την απόδοση της ενέργειας αν θέλουμε να ξεπεράσουμε την κρίση. Η ενεργειακή αποδοτικότητα και ο τομέας αυτός είναι τομέας δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης. Χρειάζονται επενδύσεις επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, κάτι που θα ενισχύσει και την κοινοτομία. Η στρατηγική και οι στόχοι της στρατηγικής 2020 ε, όσον αφορά την ε, κατανομή της βοήθειας και της στήριξης δεν θα πρέπει να αγνοήσουν τις ε, τοπικές αρχές, την τοπική αυτοδιοίκηση, περιφερειακές αρχές που θα πρέπει να έχουν καλύτερη πρόσβαση ε, στις πηγές χρηματοδότησης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συγχαρητήρια στην κυρία Κλέβε για αυτή την εξαιρετική έκθεση στην οποία επενθυμίζει ότι θα πρέπει να λάβουμε μέτρα για την ενεργειακή απόδειση, η οποία είναι απαραίτητη γιατί βοηθά την ανταγωνιστικότητα και συνεισφέρει ε, στην ενεργειακή επάρκεια. Ε, πρέπει να πούμε ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν στο μέγιστο βαθμό τα κονδύλια των διαρθρωτικών ταμείων ε, και των υπόλοιπων κονδυλίων, τα οποία είναι αφιερωμένα από Ευρωπαϊκή Σκοπιά στην ενέργεια. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν δυνατότητε σε επίπεδο προτεραιότητα, να υποστηρίξουμε τι ανανεώσιμε πηγές ενέργειας, να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στη σχέση μεταξύ ε, της ενεργειακής απόδοσης και των πιο ευάλωτων ε, χρηστών ε, και επίσης να λάβουμε υπόψη τις γεωγραφικές ιδιωτηριότητες των εξόχως απομακρυνμένων περιοχών. Για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020 θα έχουμε νέες δυνατότητες ώστε ε, τα ε, ταμεία συνοχής και τα διαρθρωτικά ταμεία να χρησιμοποιηθούν προς όφελος αυτής της καλύτερης ενεργειακής απόδοσης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η Αντιπρόεδρος Ρέντινγκ, εκ μέρους Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Κλεβακέκους ε, γιατί όσα έκανε για αυτή την έκθεση, διότι Πρόκειται για μια διεξοδικότατη έκθεση, η οποία σίγουρα θα βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει τη δράση της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί με την άποψη ότι τα μέσα της πολιτικής συνοχής θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για επενδύσεις στην ενέργεια και να συνεισφέρουν ε, στην ανταγωνιστικότητα, στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στην ανάπτυξη. Όπως είπε και η ίδια η συγχύτρια, είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, και σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο να μπορέσουμε να έχουμε συνεισφορά ώστε να επιτευχθούν οι φιλόδοξοι στόχοι του ενεργειακού τομέα, διότι οι περιφέρειες και οι πόλεις μπορούν να βρουν ε, λύσεις επιτόπου ε, όπως έχει αποδείξει το έργο των δημάρχων στο παρελθόν. Ε, το αυτό ισχύει και για τα μέτρα για την ενέργεια στα προγράμματα της πολιτικής συνοχής και είναι επίσης πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε να έχουμε και μια σειρά από πρότυπα μέσα ε, καθώς και ένα συγκεκριμένο μέσο για την εξέλιξη της ενεργειακής απόδοσης ε, στις, στα κτίρια κατοικιών στις πόλεις. Και θεωρούμε ότι θα πρέπει οι πολιτικές αυτές να ευρεωθούν καταλήλως ε, και θα προσπαθήσουμε ε, από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής να το κάνουμε αυτό. Υπάρχει και νέα οδηγία για την ενεργειακή απόδοση η οποία θα ε, φέρει πραγματικά την καινοτομία των κτηρίων στο, ε, στην πρώτη γραμμή ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους της απόδοσης για το 2020. Θα πρέπει να είναι μια πολιτική που θα προσανατολίζεται στα αποτελέσματα, γι' αυτό ακριβώς προσπαθούμε να δώσουμε πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές για το σχεδιασμό και την εφαρμογή των επενδύσεων στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης κτηρίων ε, στα πλαίσια της χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής. Θέλουμε να έχουμε το μέγιστο δυνατό βαθμό των ιδιωτικών επενδύσεων ώστε να αποτελέσουν κίνητρο για μια καλά λειτουργούσα αγορά. Ε, σε καιρό σοβαρής οικονομικής κρίσης είναι πολύ πιο σημαντικό από ποτέ να έχουμε ε, επενδύσεις με την υψηλότερη προστιθέμενη αξία. Ε, γίνονται εντατικέ προσπάθειες για τα προγράμματα των πόλεων για την επόμενη προγραμματική περίοδο και θα πρέπει όλα αυτά να τα προσερμίσουμε στις ανάγκες τους και να δούμε και τι δυνατότητε έχουν αυτέ οι περιφέρειες. Έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε μια επιτυχή λύση. Σας ευχαριστώ. Τελείωσε η συζήτηση. Η ψηφοφορία επίσης αύριο στις 12. Περνάμε στο επόμενο σημείο της μερίσιας διάταξης. Την έκθεση του κυρίου Γκουίντο Μιλάνα για την στρατηγική για την αλληλεία στην Αδριατική